κάνουμε ό,τι μπορούμε ως πολίτες για να αποφύγουμε και να, αυτά το φαινόμενο και να σώσουμε τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Πόρτας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τον λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αποτελεί συμβιβασμό ανάμεσα στις, ε, σε ομάδες με πολύ διαφορετική άποψη για τις πολιτικές επασχόλησης ε, και προστασία της ανεργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές και τις ε, Επιτροπές Απασχόλησης και Προπολογισμών γιατί μας ε, βοήθησαν να καταλήξουν αυτή τη συμφωνία που θα βοηθήσει, που θα προστατέψει αυτούς που είναι θύματα πολίσεων. Ε, δύο διαπιστώσεις. Πρώτον, οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης θα συνεχίσουν να είναι αισθητέ ακόμα και αν η ανάκαμψη γίνει πραγματικότητα. Πράγμα που έτσι κι αλλιώς τίθεται υπό αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, οι μαζικές απολύσεις δεν αποτελούν κομμάτι του παρελθόντος. Θα συνεχίσουν να σημαδεύουν την κοινωνική ζωή των χωρών μας και στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο η πρώτη επιλογή είναι απλή. Θέλουμε να επιμηκύνουμε μέχρι το 2020 την χρήση του Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Το μόνο μέσο που η Ευρώπη ε, προορίζει ε, για την αποζημίωση ε, σε απολυμμένους. Η απάντηση είναι σαφής. Ναι, θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς τους ε, ε, ανέργους. Ναι, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω ε, προγραμμάτων επανένταξης και κατάρτισης. Ναι, θέλουμε ότι αξίζουν μια καινούργια ευκαιρία και εμείς οι πολιτικοί υπεύθυνοι τους το χρωστάμε. Δεύτερη διαπίστωση. Αυτό το ταμείο, παρόλο ότι έχει πολλές αδυναμίες, βελτιώθηκε μέσω των τροποποίησεων που έγιναν στον κανονισμό του. Ε, αυξήθηκε ο αριθμός των υποψηφίων, για παράδειγμα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί, αλλά ήδη μπορούμε να εντοπίσουμε το βασικό κόλλημα. τα ανάμεσα στη στιγμή που γίνεται η μαζική απόλυση και στη στιγμή που φτάνουν τα χρήματα περνούν 12 έως 17 μήνες και μερικές φορές και ακόμα και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά η απάντηση είναι πολύ πιο επίγουσα. Η απάντηση όμως έρχεται με ταχύτητα σαλιγκαριού, χελώνας. Πολλοί εργαζόμενοι τελικά δεν καταφέρουν να επωφεληθούν αυτών των ποσών. Απ' την άλλη μεριά ε, οι καθυστερήσεις αυτές ε, αποθαρρύνουν ε, την υποβολή υποψηφιότητων σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι, πολλές φορές οι αρχές οι, οι ίδιες ε, αργούν να ε, αποζημιώσουν τους εργαζόμενους, περιμένουν να εγκριθούν οι ενισχύσεις από την ε, Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Αυτό δημιουργεί σημαντικότατα προβλήματα, ιδιαίτερα σε λιτότητα. Συνεπώ, η έκθεση προτείνει μια σειρά μέτρων βράχη πρόθεσμων για να μειωθεί κατά 50% η καθυστέρηση. Προτείνουμε το Ταμείο να γίνει μόνιμο από το 2013 και μετά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Ορισμένα από τα, τα, ε, κάποια από τα κράτη που πιο πολύ έχουν υποφεληθεί από το Ταμείο επιμένουν στην απλοποίησή του. Ε, ακριβώς για να μπορούν να ε, ζητούν, ζητήσουν περισσότερα ποσά. υπάρχει ο κίνδυνος, ο, ε, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει είτε ο, το Ταμείο είναι αργό είτε είναι γρήγορο γιατί εξαρτάται από τι επιπτώσεις της, ε, των πολιτικών λιτότητας ε, που στον προπολογισμό μας. Αυτό που συζητούμε είναι κάτι άλλο. Λέμε ποια θα είναι η στάση της Ευρώπης έναντι των μαζικών απολύσεων. Ε, θα θυσιαστούν οι εργαζόμενοι στο βωμό της, της δημοσιονομικής λιτότητας. Θα πρέπει να δώσουμε εξίσου μεγάλη προσοχή στο ε, χρηματοοικονομικό σύστημα και στους εργαζόμενους. Γιατί αυτό απορρέει από την ηθική μας, από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την Ευρώπη. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι απαραίτητα κοινωνική. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Περνάμε απευθεία στο KTI και όπως φαντάζεστε Έχουμε περισσότερες ενδιαφερομένους από ό,τι χρόνο, οπότε δεν χρειάζεται να ζητήσει άλλο τον λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μπασέσκου λοιπόν για ένα λεπτό. Να κάνω μερικά σχόλια που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εννιά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία ε, ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της ε, παγκοσμιοποίησης δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα αυτό το ταμείο. Ένας από τους λόγους είναι ο πολύ περιοριστικός χαρακτήρας των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Ακόμα και μετά την αναθεώρηση που έγινε το 2009. Το ταμείο αυτό είναι χρήσιμο υπό την προπόθεση ότι θα είναι ευέλικτο. Οι ρωμανικές ε, αρμόδιες αρχές δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα και σήμερα το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση τον πόρων αυτού του ταμείου. Εν τω μεταξύ τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρούμε αύξηση της ανεργίας ε, στη Ρουμανία και η χώρα μας ε, έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα, ε, σημαντικό πρόγραμμα ανασύστασης της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι αυτό το ταμείο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσετε και την ευκαιρία να μιλήσω. Θεωρώ πως ε, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει ζωτική σημασία και πρέπει να στηριχθεί η ανάγκη. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απολύονται χωρίς να φταίνε, να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Εγώ συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι ωφελήθηκαν από αυτό το ταμείο και αυτό βεβαίω αντανακλά τη νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι δηλαδή, ότι η νέα κυβέρνηση ζητάει να σταματήσει η λειτουργία αυτού του ταμείου. Ένα ταμείο το οποίο βοηθά τους εργαζόμενους. Ε, ελπίζω λοιπόν να επανεξετάσουν αυτή τους την στάση. Πρέπει να το στηρίξουμε, να το προστατεύσουμε και βεβαίως να γίνουν ρυθμίσεις όπου πρέπει. Πρέπει να στηρίξουμε αυτό το ταμείο και θα ήθελα να χρησιμοποιηθεί και με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Πόρτας για το έργο του. Ε, στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν δύο περιοχές στις οποίες ε, επενεύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να πω πως είναι πολύ θετικός ο ρόλος του και η Κομισιόν ήρθε και εξήγησε την λειτουργία του στους εργαζόμενους. Κάποιος το χαρακτήρισε ένα δώρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν το νόημα βέβαια, αλλά η εφαρμογή κάπως απογοήτευσε τους ανθρώπους. Νομίζω πως πρώτα απ' όλα αυτό οφείλεται στις κρατικές υπηρεσίες. Μία από τις οποίες είναι γνωστή για ε, λανθασμένη χρήση κονθυλίων στο παρελθόν στην Κομισιόν, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ δυσκίνητοι όταν προσπαθούν οι άνθρωποι βεβαίως να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση και βεβαίως όσον αφορά το χρόνο εκταμίευσης των ε, χρημάτων. Πρέπει δηλαδή να δούμε πότε ε, γίνεται η αίτηση και πότε εκταμείευε τα χρήματα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ κύριε Στάτν. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόληση και Προπολογισμού οδήγησε σε ένα πολύ καλά δομημένο σχέδιο έκθεση Χαίρομαι από όλα αυτά που ε, περιέχει και που αφορά το μέλλον του Ταμείου αυτού, όπω για παράδειγμα την απαραίτητη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για την κατάρτιση των φακέλων ή στην προσοχή που θα πρέπει να δίνεται ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εξάλλου, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μελετηθεί το θέμα της χρηματοδότησης και για το μέλλον. Ε, θα πρέπει αυτή την κοινωνική Ευρώπη την οποία θέλουμε να τη συνοδεύσουμε και με συγκεκριμένα μέσα. Ορισμένοι βεβαίω δεν βλέπουν τα πράγματα κατά από την ίδια σκοπιά. Ε, ε αυτό όμω ε, θα, ήταν, θα έπρεπε να αναφερθούν και μέσα στην ίδια την έκθεση όλε οι πιθανέ οδοί για χρηματοδότηση. Να βελτιώσουμε λοιπόν αυτό το εργαλείο και να ψηφίσουμε θετικά ε, ε, διακόπτη πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ και τελευταία στο γύρο και η κυρία Φιγκερέδο. Θέλω να υπογραμμίσω τρία ακόμα ζητήματα σχετικά. Πρώτον, μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να ληφθούν για να παρεμποδιστούν οι μετακινήσεις πολυεθνικών εταιριών και να καταπολεμήσουμε έτσι την ανεργία. Δεύτερον, η εφαρμογή αυτού του ταμείου, η χρήση του, που δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να διευκολυνθούν αιτιολογημένες ε, απολύσεις ε, λόγω μετακινήσεων πολυεθνικών ή λόγω αναδιαρθώσεων τους. Τρίτον, να υπογραμμίσω την ανάγκη αύξησης της ε, κοινοτικής συμμετοχής από το 65% σε ένα μίνιμουμ 80% έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσφυγή στο Ταμείο εκ μέρους ε, κρατών μελών που έχουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα και ε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που πιο πολύ το χρειάζονται να υποστηριχθούν το συντομότερο δυνατό. Κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος ο κ. Σιόλος εξ ονόματος Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον κύριο Πόρτα, τον εισηγητή, για την εξαιρετική του αυτή εργασία που οδήγησε σε αυτή την πληρέστατη έκθεση. Ε, μέσα από συνεργασία βεβαίως και με τους ε, ε, εκπροσώπους των άλλων επιτροπών ε, αυτή η έκθεση έρχεται την κατάλληλη στιγμή γιατί θα συμπεριληφθεί χωρί πρόβλημα στην εργασία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, γιατί έχουμε ορισμένα συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα. Πρώτα απ' όλα, παρέκκληση. Ε, λόγω κρίσης για να αντιμετωπίσουμε τους απολυμμένους λόγω της οικονομικής ε, και χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και για χρηματοδότηση 67% που λύγει το 2011. Εδώ θα πρέπει να δούμε κατά πόσα μπορούμε να παρατείνουμε την ε, παρέκκληση αυτή ή να ε, επανέλθουμε στι απολύσει με ε, ποσοστό χρηματοδότηση 50%. Δεύτερον, δεύτερο χρονοδιάγραμμα, τέλο του 2013, εκεί όπου όλοι οι κανονισμοί του ΦΕΜ, ε, του Ταμείου, θα πρέπει να επανεξεταστούν. Και ένα από τα ζητήματα είναι το κατά πόσον τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα επόμενα, στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η έκθεση του κ. Πόρτα υποστηρίζει τους ίδιους τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του Ταμείου και τονίζει την αναγκαιότητα ε, συνέχισης της ζωής του Ταμείου αυτού. Ε, πράγματι, ε, αυτή αποτελεί μία από τις επιλογές ε, στο μέλλον και η συγκεκριμένη έκθεση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει την επιλογή αυτή. Η έκθεση Πόρτας προτείνει ενδιάμεση αναθεώρηση που προβλέπεται στο 2011 να ολοκληρωθεί μέχρι την 30 Ιουνίου του 2011. Κοιτάξτε, αυτό έχει προβλήματα σε σχέση με τον κανονισμό του Ταμείου, διότι η έκθεση όσον αφορά την πρώτη ε, οι εκθέσει για τι πρώτε υποθέσει που θα έχουν εξεταστεί ε, μετά από την αναθεώρηση του κανονισμού για το Ταμείο θα είναι έτοιμε τον Νοέμβριο 2011. Και ε, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να δούμε τι γίνεται με τον κανονισμό. Να δούμε, για παράδειγμα, το ποσοστό επιτυχία των δράσεων του Ταμείου, να υπάρξει συγκριτική ανάλυση των μέτρων, να υπάρξει διαδικασία διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου και ανάλυση των επιπτώσεων του Ταμείου επί των δικαιούθων. Η, η, η έκθεση αναφέρει ότι μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα ήταν μάλλον ε, παθή Ε, υπολογίζοντας ότι ε, ε, μόλις εννέα κρατημέλη εκπροσωπούνται ε, στη δράση αυτή με την έννοια ότι ε, υπήρξαν, όχι συγγνώμη, εννέα κράτη-μέλη δεν έκαναν κανένα, δεν υπέβαλαν κανένα αίτημα και υπήρξε ε, υποχρησιμοποίηση των κονδυλίων που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν όσον αφορά τα 11 πρώτα, τα 11 πρώτα αιτήματα. Ε, και ζήτησε η Επιτροπή επιστροφή περίπου του 40% των ποσών. Υποστηρίζω, όπω αναφέρει και η ίδια έκθεση, ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν ε, τι υποθέσει που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του αρχικού κανονισμού. Γιατί, όπω πολύ σωστά αναφέρει και η έκθεση, η τροποποίηση του κανονισμού οδήγησε σημαντική αύξηση των αιτήσεων ενίσχυση ε, στα πλαίσια του Ταμείου αυτού όσον αφορά συγκεκριμένε ε, δράσει. Η έκθεση, πολύ σωστά, ζητά να υπάρξουν βελτιώσει, κυρίω όσον αφορά τη μείωση τη ε, διάρκεια τη διαδικασία από την απόλυση μέχρι την καταβολή των κονδυλίων από το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή. Ορισμένε όμω βελτιώσει από αυτέ που αναφέρονται θα ε, απαιτήσουν καλύτερη οργάνωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ε, της, ε, των δημοσιονομικών αρχών, τη Επιτροπή και των κρατών μελών. Στενή συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, με το Κοινοβούλιο, κυρίω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η στενή συνεργασία θα επιτρέψει να μειωθεί μέρο τη καθυστέρηση αυτή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλουν αιτήματα μόλι ανακοινώνονται οι απολύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μεριά τη θα πρέπει να παρέχει ε, τι ε, αναγκαίε πληροφορίε και συμβουλή στα κράτη-μέλη και να ορίζει ένα χρονικό διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών για την αξιολόγηση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, σημειώνουμε την παράταση τη παρέκκληση για την κρίση μέχρι το δημοσιονομικό πολιτέ πλαίσιο. Κοιτάξτε, μέχρι το 2013 θα έχουν εξεταστεί απόλυτα τα σημεία αυτά στα πλαίσια ε, των προετοιμασιών για διαπραγμάτευση του δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου και σίγουρα μέρος της, ε, ε, των επιλογών είναι και η επιλογή που αναφέρεται μέσα στην έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και άλλωστε προβλέπεται μία σειρά διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη και με τους άλλους ενδιαφερόμενους και είμαι σίγουρος για το ότι οι εισηγητές αλλά και ο εισηγητή ε, και οι υπόλοιποι, ε, τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου, θα συμβάλλουν επικοδομητικά στι ε, διαπραγματεύσει αυτέ, γιατί στόχο είναι να βελτιωθεί το μέσο και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό στο μέλλον, διότι είναι ένα μέσο το οποίο αποδεικνύει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στου εργαζόμενου που απολύονται. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Άρα τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση. Η ψηφοφορία είναι αύριο στι 12.30. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακολουθεί τώρα η έκθεση του κυρίου Λέχνερ, διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων και τον λόγο έχει ο εισηγητής για 4 λεπτά. Ευχαριστώ.